συνάδελφο Μάρκ Ιώζεφ Γκορμπάτσεκ και Ντάβιτ Μπόνταν Γιαβιέτσιτς ε, διορίστηκαν μέλη της πολωνικής κυβέρνησης. Ε, συγχαίρω λοιπόν τους συναδέλφους ε, για την ανάληψη αυτού του αξιώματός τους και έτσι λοιπόν το Κοινοβούλιο διαπιστώνει το ότι από τις 16 Νοεμβρίου και μέχρι σήμερα χειρεύει η θέση αυτών των δύο